Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Καταρχήν για την έκθεση Στίβενσον. Κυρία Τσανίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός του Συμβουλίου για το Πολιετές Πρόγραμμα για το απόθεμα Ρέγκας εγκρίθηκε πριν τη θέση σε ίσχυ της ε, συνθήκης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει ευθυγράμμιση. Ο κανονισμός αυτό, ο πρώτος στο τομέα της αλίας, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη επειδή θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Η λύση που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που ισχύει για άλλα πολιετή προγράμματα. Γι' αυτό, λοιπόν ακριβώς το λόγο υπερψήφισα την πρόταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Τσανίκη. Συνάδελφος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι το περιεχόμενό της και όσον αφορά το περιεχόμενο δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση γιατί και βέβαια είναι σημαντικό να παρακολουθούμε το απόθεμα ρέγκας και την υπερβολική αλίευση και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά και το άλλο τμήμα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό υποστηρίζω αυτή την έκθεση μεταξύ άλλων. Είναι το θέμα του τι κάνουμε με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πότε έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξεις και πότε έχουμε μία συνήθη νομοθετική διαδικασία και εγώ υποστηρίζω σαφώς την ε, πρόταση του εισηγητού ότι θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, γιατί θέλουμε να έχει την πολιτική εξουσία το Κοινοβούλιο και γι' αυτό είμαι της γνώμης ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει εύκολα να ε, χωρεί εξουσιοδοτή στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Συνάδελφος Κέλλη. <coughs> Uh, Κύριε Πρόεδρε, άκουσα όλη τη συζήτηση που διεξήχθη σήμερα το πρωί στο ημικύκλιο για την έκθεση Στίβενς και μου προξένησε αποτροπιασμό το ότι δεν αναγνωρίζεται δεν γίνεται σεβαστή η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να κατανοήσουμε τότε ο Πάτε Κόπο και άλλοι και ο κ. Στίβεν, προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν ούτω ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα του αλληλευτικού κλάδου. Αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί. Είναι αδικία. Είναι απαράδεκτο. Οι περισσότεροι ψηφίσαμε υπέρ της εκθεσής 500 95 από του 610 ψήφισαν υπέρ. Ελπίζω ότι αυτό θα δώσει κίνητρο. Και ο κύριος Στίβενσον θα συνεχίσει την προσπάθειά του. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Κύριος Καμάλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία που μας δίνετε θα σας εξηγήσουμε τι ψηφίσαμε. Συγχαρητήρια προς τον κύριο Στίβενσον που ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσπαθειά του. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η κοινή πολιτική ε, έχει αποτύχει. Ε, θα μπορούσε να είναι κομμουνιστική πολιτική, κεντροκατευθυνόμενη, ε, διότι τελικά είναι μη βιώσιμη πολιτική, πρόκειται για, για ψάρεμα σε θαλάσσες που δεν έχουν ψάρια. Θα έπρεπε όμως να ρίξουν μια ματιά την Ισλανδία, την Νέα τα νησιά Φόκλαντ, που είναι παραδείγματα προς μίμηση σε σχέση με το πώς ρυθμίζουν τα δικαιώματα που υπάρχουν, την κληροδότηση αυτών κλπ. κλπ. Από οικογένεια σε οικογένεια. Και έτσι οι αληθικοί πόροι διατηρούνται. Δεν υπάρχει αυτού του είδου η κεντροκατευθυνόμενη κομμουνιστική διαχείριση. Έτσι άδειασαν από ψάρια οι θάλασσές μας. Θα έπρεπε να, είναι, ε, να έχουμε μια προσέγγιση αγοράς. Ευχαριστούμε κύριε Καμάλη. Ο κύριο Τάνοκ. κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ ε, σε σχέση με, αυτή την ε, ε, έκθεση για τη Ρέγκα Δυτικά τη Σκοτία. Νομίζω ότι θα πρέπει οι διεθνεί φορεί να βοηθούν περισσότερο να βάλουν υπόψη και έτσι θα πρέπει το, το, Συμβούλιο για τα Παλαιτικά Είδη ε, και η Επιστημονική Επιτροπή για την Ελία θα έπρεπε να έχουν γνωμοδοτήσει πριν γίνουν αλλαγέ στο πολιτέ πρόγραμμα. Θα πρέπει έτσι να φροντίσουν τη διατήρηση των πόρων, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη, τα, τους, νεογνούς και θα έπρεπε να έχουμε πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες ρυθμίσεις και έτσι να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ελευτικών πόρων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ωραία. Ολοκληρώθηκαν οι επεξήγησει ψήφου για αυτή την πρώτη έκθεση Στίβενσον και τώρα για την έκθεση Άντερη, η κυρία Τζανίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι Μποπάλ της ε, Τουλούζης και τόσες άλλες εταιρείε ε, που έχουν ε, θέσει σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Το κείμενο του συναδέλφου Άντερ έχει να κάνει με την οδηγία σε Βέζο 2 που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει ατυχήματα που αφορούν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που μπορεί να έχουν ε, διαχειριστεί στο περιβάλλον. Από τον Ιούνιο του 2015 θα έπρεπε να ληφθούν τα μέτρα για να προληφθούν ακριβώς αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Τσανίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουμε γνωρίσει μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι είναι πολλές περιπτώσεις όπου τα εργατικά ατυχήματα συνοδεύονται και από καταστρεπτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι κινδυνεύει η υγεία των πολιτών και όχι μόνο μίας χώρας κάθε φορά. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υποκατασταθεί η οδηγία 96, γι' αυτό υποστηρίξα την πρόταση του συναδέλφου, ώστε ακριβώς τα επίπεδα σημερινή προστασία όχι απλώς να διατηρηθούν, αλλά να ενισχυθούν περαιτέρω. Πιστεύω επιπλέον ότι οι νέε διατάξει θα πρέπει να είναι σαφέστερε, συνεπέστερε και να διευκολύνουν την κατανόηση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ε, ευέλικτε τι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας για να μπορούμε να ε, τροποποιήσουμε και το παράρτημα Ή, εφόσον υπάρχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες από την ευθυγράμμιση με τον κανονισμό 1267. 62. Και επειδή μπορεί να υπάρξει αντίτυπος ε, στις επικίνδυνες ουσίες. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνιώτση. Συνάδελφος Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ψήφισα υπέρ αυτής της εκθέσεως, διότι στην περίπτωση τέτοιων μεγάλων ατυχημάτων θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση του κοινού. Θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τις αιτίε αλλά και τις συνέπειες αυτών των ατυχημάτων δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο από τέτοιου είδου ατυχήματα για το πόσο επικίνδυνο είναι για την δημοσία υγεία. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηροί. Και η ενημέρωση του κοινού να γίνεται πιο ολοκληρωμένη. Νομίζουμε ότι με αυτή την έκθεση θα βοηθήσουμε στο να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Γιάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ατυχήματα στο παρελθόν, όπως στο Σεβέζο, που χτίσαν τη ζωή πολλών ανθρώπων, έδειξαν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα και πώς πρέπει να προλαμβάνουμε με προληπτικά μέτρα για να μην συμβαίνουν μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες. Πρέπει να έχουμε λοιπόν τα κατάλληλα μέτρα στη διάθεσή μας και γι' αυτό είχαμε τις οδηγίες σε Βέζο 1, σε Βέζο 2 και τώρα τη Σεβέζο 3 και είναι υποχρεωμένες οι αρχές και στα κράτη-μέλη να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν ατυχήματα και υπάρχει μια προσέγγιση πολλαπλών σταδίων για να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να, ε, εφαρμόζεται, ε, να εφαρμόζονται σχέδια εκένωσης και σχέδια πρόληψης στους χώρους όπου αυτό απαιτείται. Αυτό δείχνει πόσο ε, σημαντικό είναι αυτό ο τομέας και γι' αυτό υποστήριξα αυτή την ε, έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιάρ, συνάδελφος Άνναν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεδομένου των όσων συμβαίνουν εκτός αυτής της αίθουσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, εμείς να περνάμε τόσο χρόνο μιλώντας για μεγάλα ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες. Νομίζω ότι φαίνεται ότι υπάρχει κάτι πολύ ζωφερό στην εκτασία αυτή, διότι η πιο επικίνδυνη ουσία από όλε φαίνεται να ήταν το ευρώ. Δεν το εννοώ κυριολεκτικά. Καταλαβαίνω ότι μερικοί έχουν αλλεργικέ ε, αντιδράσει και σε άλλε ουσίε, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Ένα θέμα, μια ευκαιρία να συζητήσουμε κατά του κοινού νομίσματο. Όμω, πώ παρασύρθηκαν τόσο πολύ από το όραμα τη Πολιτική Ένωση οι ηγέτε μα, ε, ξεχνώντα του οικονομικού κινδύνου που, κινδύνους που μπορεί να προκύψουν μαζί με τι ε, καταστρεπτικέ συνέπειε που βλέπουμε γύρω μα σήμερα. Ένδια, την ε, υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, τη μετανάστευση, όλα αυτά γιατί, γιατί τόσο πολύ είχαμε αγαπήσει αυτό το όνειρο τη στενότερη ένωση. Εκτό του κοινοβουλίου τη Βρυξέλλε υπάρχει ένα άγαλμα μια θηλυκή μορφή που κρατά το ευρώ. Ε, μια γυναίκα μάλλον που κρατά ένα νόμισμα, το ευρώ ω σύμβολο. Κατά τα άλλα όμω. Πραγματικά νομίζω ότι γύρω από αυτό επικρατεί καταστροφή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χανον. Σας ακούμε παρότι μιλάτε εκτός θέματος. Συνάδελφος Μπασέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτή τη εκθέσεω, διότι η πιθανότητα για τέτοιου ατυχήματα θα πρέπει να περισταλεί στην ε, Ουγγαρία στο Match Light το 2010. Ήταν μια τέτοια περίπτωση που δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να περιορίσουμε τη ζημία προς το περιβάλλον και προς τον κόσμο. Νομίζω ότι η οδηγία λειτουργεί καλά. Όμως θα πρέπει να τροποποιηθεί και έτσι να βελτιώσουμε την εφαρμογή της και θα πρέπει να μειωθεί το διοικητικό βάρος. Επίσης, ε, οι πιο σημαντικές τροποποίησεις θα πρέπει να αφορούν την πρόταση στην ενημέρωση και την συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία χρειάζεται. Και η οδηγία επομένω καθ' τον τρόπο θα πρέπει να υποστηρίξει τροποποιήσει. Η πρόσβαση επίση στη δικαιοσύνη θα πρέπει να βελτιωθεί και νομίζω ότι η ενημέρωση του κοινού είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έτσι έχουμε κλίμα εμπιστοσύνη. Όταν ο κόσμο έχει ασφαλεί και ακριβεί πληροφορίε, τότε μπορούν να λάβουν τα σωστά μέτρα σε περίπτωση ατυχήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Καμάλ. Thank Καμάλ, ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη το τι γίνεται και με τα τοξικά υλικά και είναι σωστό ότι γι' αυτό ελήφθη υπόψη στα πλαίσια της μετώπιση αυτής τη κατάστασης είναι επίσης ε, σημαντικό. Για να δούμε τι γίνεται επίση και με το τοξικό χρέο μια που τόσε κυβερνήσει δαπανούν πολύ περισσότερο από όσα θα έπρεπε, από όσα θα μπορούσαν. Τοξικό χρέο. Πιο πολλά είναι τα έξοδά τους από τα έσοδά του και τελικά στριμώχνονται να δούμε τι γίνεται και αυτό το, το, το, το, την ηθική διακινδύνευση, το moral hazard όσον αφορά το τι γίνεται με τις τράπεζες. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να φερθούν πιο υπεύθυνε σχέση με τι καταθέσει. Και είδαμε πόσο κινδυνεύουν κάποιε χώρε που δεν είναι ανταγωνιστικέ από το ευρώ. Είδατε τι έπαθε η Ελλάδα και η Ισπανία. Δεν μπορούν. Άρα θα πρέπει όλες αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις και αιτίε να τις αντιμετωπίσουμε που καταντούν επέντε στις χώρες. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμάλ. Τάνοκ. Όχι, όχι, λάθο. Ήταν για άλλη έκθεση. Οπότε ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Άντερ και περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση ΡΙΣ. Συνάδελφο Αντωνιώτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία 2009 της 6 η Μαΐου 2009 δηλαδή για τα τρόφιμα που προορίζονται για τη διτροφή βρεφών και παιδιών ορίζει τις γενικές διατάξεις που θα καθορίζουν τη σύσταση και την σύνθεση τέτοιων τροφίμων. Οι διατάξεις της οδηγίας βεβαίως ανταποκρίνονται κυρίως στα πορίσματα του 1977. Δεν καλύπτουν τι σημερινέ καταναλωτικέ ανάγκε, γι' αυτό χρειαζόταν αυτή η ε, ριζική αναθεώρηση τη οδηγία και γι' αυτό και υπερψήφισα την πρόταση τη συναδέλφου Ρή. Θεωρώ παρά όλα αυτά αναγκαίο να προστατεύσουμε περισσότερο του καταναλωτέ, να απλουστεύσουμε την νομοθεσία και γενικότερα να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε που τα κράτη-μέλη και οι φορεί ε, του τομέα αυτού αντιμετωπίζουν στο να ε, υλοποιήσουν τι ισχύουσε νομοθετικέ διτάξει σε όλα τα διατροφικά ζητήματα. Θα έπρεπε με ενιαίο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχουν παρόμοιε προποθέσει για όλου του ε, εμπορευόμενου στον τομέα αυτό, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και του τελικού καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ προσπάθησα να ψηφίσω υπέρ αυτής της εκθέσεως, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργήσε. χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση όπως προβλέπει αυτή η έκθεση και στοχεύουμε στο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ανηλίκους. Η επαχυσαρκία των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Και φυσικά και οι διαφημίσεις επηρεάζουν τον τρόπο διατροφής των ανηλίκων. Είναι ξεκάθαρο ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες. Εγώ συμφώνησα με τα όσα προτείνονται εδώ γιατί η διαφήμιση δεν έχει ως σκοπό την ενημέρωση αλλά την κερδοφορία. Πολλές φορές επομένως είναι τελείως ασυνείδητοι οι διαφημιστές. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να κερδίζουν με προϊόντα γεμάτα ζάχαρη και λύπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον Ιούνιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει μια πρόταση και συγκεκριμένε στη συνέχεια διατάξει ε, για τα είδη διατροφή ε, που προείζονται για ειδικού ιατρικού σκοπού. Υπάρχουν ε, όλα αυτά τα οποία μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα θετικά, αλλά στην πράξη να εμφανίζονται ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που πρέπει να τηρήσουν συγκεκριμένε δίαιτε και χρειάζονται συγκεκριμένα συστατικά και γι' αυτό είναι ευγνώμων προ την Επιτροπή Περιβάλλοντο Δημόσια Υγεία που επέλεξαν αυτό αυτό το αντιφατικό θέμα. Χρειαζόμαστε επαρκείς πληροφορίες ε, ε, που να μην μας κατακλείζουν όμως και να μην υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν ε, που υπάρχει αυτή η έκθεση για να μπορέσουν και στην πράξη να εφαρμοστούν αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τόσους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εγώ ψήφισα υπέρ της εκθέσεως. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές τις οποίες ψήφισαμε σήμερα. Τροπολογούμε έτσι την οδηγία του 1974, αλλά επίσης προστίθεται εδώ η προστασία κάποιων ευάλωτων κατηγοριών πολιτών. Πολύ σημαντικό. Πολλές φορές πέφτουν θύματα παραπλανητικής ετικετοθεσίας οι πολίτες. Και πολλές φορές έχουμε και δυσκολίες στη ιατρική αγωγή που να τους παρουσιάσουμε μετά, ας πούμε την δυσανεξία στην γλουτένη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχητικά επίπεδα της ε, λεγόμενης κοιλιακής ασθενείας στην Ευρώπη της ορθότερα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και συνδετικά μέτρα και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστούμε. Τα ράφια, του σούπερ μάρκετ, τα ράφια των σούπερ μάρκετ μάλλον είναι γεμάτα από τρόφιμα τα οποία υποτίθεται ότι καλύπτουν συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες για ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος, για αυτούς που θέλουν να κερδίσουν βάρος. Θα πρέπει λοιπόν οι καταναλωτέ να έχουν την επιλογή, αλλά να καταλαβαίνουν και να κατανοούν τι αγοράζουν και καταναλώνουν. Η έκθεση αυτή απαιτεί σαφέστερου και παρόμοιου κανόνε για την αντικειτοθεσία σε διαιτητικά προϊόντα. Εδώ τα κράτη-μέλη, όταν θελοποιούν την νομοθεσία αυτή, θα μειώσουν παρά θα αυξήσουν ε, τα απαγορευτικά όρια, την γραφειοκρατία μάλλον. Θα πρέπει εδώ να διευκολύνουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Οι καταναλωτές χρειάζονται σαφείς οδηγίες και απλούς κανόνες οι εταιρείε ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Για τους λόγους αυτούς στήριξα την έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Γιανακουδάκη. Συνάδελφος Τάκουλα. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση ΡΙΣ και συγχαίρω την κυρία ΡΙΣ για το εξαιρετικό αυτό κείμενο. Όταν μιλάμε για ε, τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, δεν θα πρέπει να δίνουμε την εικόνα, ε, μια εικόνα διαστρεβλωμένη, διότι αυτό ακριβώς πετυχαίνει η έκθεση. Όταν μιλάμε για την κοιλιοκάκη, μας λέει πολύ ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική ιατρική αγωγή. Θα πρέπει λοιπόν όντως να επικαιροποιηθεί η σχετική νομοθεσία και αυτά τα νέα είναι πραγματικά θετικά. Έχει καταντήσει απαρχαιωμένη η ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει λοιπόν να την αναθεωρήσουμε και είναι πολύ καλό αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την εισηγητή, την εισηγητρία για την, προσέγγιση της. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η τωρινή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι ο θυλασμός είναι θετικός για τα παιδιά και ότι από τους έξι μήνες και μετά χρειάζονται διαφοροποιημένη διατροφή. Η τροπολογία 6 ε, μιλάει για την ε, μείωση της διαφήμισης όσον αφορά τα βρεφικά γάλακτα ε, να μην ε, υπάρχει σε ε, περιοδικά για γονείς που αφορούν τα παιδιά. Αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικό γιατί περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών. Θα οδηγηθούμε και στην απαγόρευση της τηλεοπτικής διαφήμισης. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των βρεφικών γαλάκτων και του γάλακτος που είναι για μετά την ηλικία του βρεφικού γάλακτος, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αποφασίζουν αν θα αποφασιστεί περαιτέρω η διαφήμιση και νομίζω ότι μια απαγόρευση της διαφήμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την εξαίρεση των συγκεκριμένων περιοδικών νομίζω ότι είναι δυσανάλογη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι διατάξει που αφορούν την ετικετοθεσία ως τα τρόφιμα για τους ε, ανηλίκους ε, όπως επίσης και τα τρόφιμα που ε, πρέπει να λαμβάνονται για ιατρικούς λόγους θα πρέπει να ρυθμιστούν όσο γίνεται καλύτερα για να προστατεύσουμε τη δημοσία υγεία και το θέμα δεν είναι το αν θα έχει ή δεν θα έχει ο κόσμος επιλογές. Απλώς θα πρέπει επιλογές να γίνονται βάσει ακριβών Άρα και η διαφήμιση θα πρέπει να διέπεται από αυστηρό κώδικα διοντολογίας και κάτι το οποίο είναι και υπέρ της βιομηχανίας. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ της εκθέσεως, διότι θεωρώ ότι η αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς είναι κάτι το πάρα πολύ εύστοχο και έτσι θα έχουμε εξορθολογισμό και στην ετικετοθεσία. Γιατί υπάρχουν κάποιες ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών. Θα πρέπει να προστατευτούν και να υπάρχει ασφαλή δικαίωση και στην προστασία του. Χρειάζεται να υπάρχει λιγότερο ιδιωτικό κόστο επίση. Και ισότητα μεταχείριση για όλα αυτά τα προϊόντα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι να υπάρχουν ισχυροί ανταγωνισμού. Μόνο χαίρετο θα έχει η ενιαία αγορά από αυτή τη ρύθμιση. Ευχαριστούμε κυρία Μπασέσκου. Ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση ΡΙΣ και το έχουμε τις προτάσεις ψηφίσματος, δημόσιες διαβουλεύσεις και διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε με τον συνάδελφο Μπίλαν. Μπίλαν, ευχαριστώ πρόεδρε Η γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ως προς την επικοινωνία, την μετάδοση των πληροφοριών και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το να διασφαλίζουμε σε όλους πρόσβαση στις δημόσιες διαβουλεύσεις στην ίδια γλώσσα είναι ανεκτήμητης αξίας ε, εργαλείο. Είναι προϋπόθεση για την ε, αρμονική συνύπαρξη στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι ένας τρόπος επικοδομητικός ώστε να ενθαρρύνουμε τον κοινωνικό διάλογο και την συμμετοχή στα κοινά. Του χρόνου θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Θα επιτρέψουμε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναλάβουν δράση σε αυτόν τον τομέα και θα επιτρέψει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες διαβουλεύσεις στη δική τους γλώσσα. Ευχαριστούμε ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δικαίωμα του κάθε πολίτου να μπορέσει να συνομιλήσει, να έρθει σε επαφή με τις θεσμικές αρχές των Βρυξελών στη γλώσσα του είναι ένα από τα ε, τελευταία προνομία πέραν της ενίας πολιτικής και πολλές φορές ως επιχείρημα στην πατρίδα μου μου λένε τι, κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι, τι, τι κάνει το Κοινοβούλιο. Ε, δουλεύει σε αγγλικά, αγγλικά, γερμανικά, αλλιώς Έτσι δεν χρειάζεται να κάνει ε, μετάφραση σε όλες τις γλώσσες ε, και ταυτόχρονα να οδηγείται σε ένα τέτοιο υπερκράτος διότι για αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο κάνουμε είναι να έχουμε τελικά μια κοινή γλώσσα στην οποία και συζητούμε όλα αυτά τα ζητήματα εδώ στο Λομέλιο γιατί αυτές οι φράσεις που δεν χρησιμοποιούμε μόνο εδώ ακούγονται σεβασμός, αναλογικότητας, επικουρικότητας πιο κοντά στον κόσμο περισσότερη, όχι λιγότερη Ευρώπη όλες αυτές οι φράσεις μόνο εδώ ακούγονται από ευρωβουλευτές και ευρωκράτες να, το είχε πει και ο Γιώργος το 1984 που είχε πει ότι μιλάει ο Λάριγκας και δεν μιλάει ο εγκέφαλος, σαν τις πάπιες. Έτσι, κλισέ. Σκέφτεται κανείς κλισέ, μιλάει με κλισέ. Γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ που βρισκόμαστε. Ευχαριστούμε κύριε Χάνεν. Κύριο Στάκουλα. Πρόεδρε, Είναι πολύ σημαντικό το ψήφισμα αυτό, γι' αυτό και το υπερψήφισα. διότι αφορά τι δημόσιε διαβουλεύσει και τη διαθεσιμότητά του σε όλε τι γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι αξιόπιστη στα μάτια των πολιτών, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίε στη γλώσσα ακριβώ αυτή των πολιτών. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Αυτό ο τομέα είναι από εκείνου όπου πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερε προσπάθειε, ώστε να έχουν όλοι οι πολίτε σαφεί πληροφορίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο των θεσμικών οργάνων, τι ενεργέ τη, όλα τα έγγραφα, όλε οι δημόσιε διαβουλεύσει πρέπει να διατίθενται σε όλε τι γλώσσε. Αυτό είναι πραγματικά θεμέλιος λήθος για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ως δημοκρατικό λοιπόν σώμα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών στην πρόσβασή τους στην πληροφορία στη δική τους γλώσσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ για να προσθέσουμε και άλλο ένα στερεότυπο στο μακρύ κατάλογο. Πολλέ φορέ μιλάμε για το δημοκρατικό έλλειμμα στο Κοινοβούλιο. Όμω, ε, πώ θα αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα. Εγώ λέω στου πολίτε ότι δεν ψηφίζεται απλώ του ε, ε, βουλευτέ, αλλά πρέπει να συμμετέχετε με όλου του δυνατού τρόπου και στη διαδικασία των δημοσίων διαβουλεύσεων. Εγώ συχνά ενημερώνω του πολίτε για τι σε εξέλιξη διαδικασίε διαβούλευση. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά σημαντικό είναι και να μπορούν οι πολίτε να επικοινωνούν στη δική του γλώσσα. Λόγου χάρη, είναι σημαντικό οι Ιρλανδόφωνοι να μπορούν να επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εθνική του γλώσσα. Όμω, η γλώσσα δεν είναι απαραίτητο ο μόνο φραγμό. Είναι εξίσου σημαντικό και τα άτομα με ειδικέ ανάγκε να επικοινωνούν με μια αποδεκτή μορφή. Νομίζω επίση πρέπει να δούμε τα χρονικά όρια. Ε, αν κανεί ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα πίεση ή σε ένα, μια μη κυβερνητική οργάνωση, είναι απλό να συμμετέχει στι διαβουλεύσει. Όμω όσοι δεν έχουν ανάλογο πόρου στη διάθεσή του, οι περίοδοι διαβουλεύσεων θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερε. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Κυρία Τζαμπόρσκα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Σε μια εποχή που όλοι και ιδίως οι πολιτικοί προσπαθούν να βρεθεί κάποιος τρόπος διεξόδου από την οικονομική κρίση, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η γλωσσική πολυμορφία έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά συνδέονται στενά αυτά τα δύο για να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει οι πολίτες να έχουν την αίσθηση του ότι ανήκουν σε ένα κοινό φορέα. Αν ε, οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν τις γλώσσες της Ευρώπης, δεν θα ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, δεν θα ενδιαφέρονται για το κοινό τους νόμισμα και το κοινό τους μέλλον. Γι' αυτό είναι τώρα περισσότερο σημαντικό από ότι στο παρελθόν να επικοινωνεί με τους πολίτες σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι πολλές δημόσιες διαβουλεύσεις γίνονται για θέματα πολύ σημαντικά και λίγοι σχετικά συμμετέχουν. Με κυβερνικές οργανώσεις, συνδικάτα και τα ΜΜΕ θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο και όλοι θα πρέπει να μπορούν εκεί να συμμετάσχουν. Αυτό θα πει η δημοκρατία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τέτοιες τάσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα πολυγλωσσίας. Και έτσι όλοι οι πολίτες Ένωση μπορούν να εμπλακούν. Σήμερα οι δημόσιες διαβλέψεις δεν έχουν οργανωθεί όπως πρέπει. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα δικαιώματα που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα για να μειώσει αυτό το έλλειμμα πληροφόρησης. Ο κύριος Τάνοκ. Εγώ απέσχουν για αυτό το θέμα των δημόσιων διαβουλεύσεων και τη διαθεσιμότητά του σε όλε τι γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια είναι σημαντικό να μπορούν όλοι οι πολίτε να έρχονται σε επαφή με τα ευρωπαϊκά όργανα στι επίσημε γλώσσε. Και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε. Και όλε οι διαβουλεύσει θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση και να είναι προσβάσιμε. Αλλά δεν υποστηρίζω το πολύγλωσσο σύστημα στα θεσμικά όργανα, διότι είναι πάρα πολύ δαπανηρό και μη αποτελεσματικό τρεις γλώσσες εργασίας, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πιστεύω ότι αρκούν. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μόνο έξι γλώσσες εργασίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης με 47 μέλη έχει μόνο δύο γλώσσες εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εποχή λιτότητας και περικοπών επιμένει ακόμη στις 23 γλώσσες. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε Τάνοκ. Ολοκληρώσαμε τις επεξηγήσεις ψήφου για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και ακολουθεί η πρώτη ψηφίσματος για την κατάσταση στο Θιβέτ. Ο συνάδελφος Χάναν ξεκινάει. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω με την αναφορά μου στο 1984. Γνωρίζουμε όλοι τη δυνατότητα της διπλής σκέψεις. Δηλαδή ταυτόχρονα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε στη σκέψη μας αντιφατικές ιδέες. Πολλοί είναι αυτοί που επιθετικά θα ήταν υπέρ των ηθαγενών και των δικαιωμάτων τους σε φτωχές χώρες του κόσμου, αλλά το ίδιο βία θα ήταν υπέρ και της μετανάστευσης και του πολυπολιτισμικότητας σε άλλα μέρη του κόσμου. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Όμως το Θιβέτ είναι μια ιδιαίτερη χαρακτηριστικότατη περίπτωση, διότι στην αίθουσα αυτή μας αρέσει να ε, συγχαίρουμε τους εαυτούς μας για το πώς ε, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, τον αυτοκαθορισμό των λαών, τα δικαιώματά τους, όμως ε, και πάλι υπάρχει εδώ η διπλή σκέψη. Διότι εάν οι Θηβετιανοί ήταν σε καλύτερη κατάσταση, αν ζούσαν με τους δικούς τους νόμου, γιατί αυτό να μην ισχύει για του Πορτογάλου, του Γερμανού και οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική κοινότητα στην Ευρώπη. Πόσο εξαιρετικό είναι αυτό να έχουμε αναπτύξει την ιδέα του εθνικού αυτοκαθορισμού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εδώ, στη δική μα την Ήπειρο, από όπου προερχόμαστε, να γυρνάμε την πλάτη στην ιδέα αυτή. Ευχαριστούμε, συνάδελφο Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού, διότι πρόκειται για μια λυπηρή πρόκληση ε, κατά της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί της Κίνας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι θετικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι παραπλανείται. Προσπαθεί να ακολουθήσει ένα αποσχιστικό λόμπι, μια ομάδα πίεσης του, του Θιβέτ με στόχο να παρενοχληθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας. Ευχαριστούμε κύριε Μπιουτικόφερο, συνάδελφος Τάνοκ. Ψήφισα υπέρ τη πρόταση ψηφίσματο για το Θιβέτ. Η κατάσταση στο Θιβέτ είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Είναι πολλά ε, τα θύματα αυτοπυρπολίσεων, μοναχοί και άλλοι και πολλά παραμένουν άγνωστα. Χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερε προσπάθειε για την αντιμετώπιση του προβλήματο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο του διαλόγου με την Κίνα θα πρέπει οι κινέζικε αρχέ να συνεχίσουν και να εντείνουν τι συζητήσει του με εκπροσώπου του Δαλάη Λάμα για την κατάσταση στο Θιβέτ πρέπει να βρεθεί μια κατάσταση που θα σέβεται την πολιτιστική διαφορά και την ύπαρξη του Θιβέτ μέσα στην Κίνα. Και η μεταφορά και άλλων κοινών υπηκών στο Θιβέτ απλώς θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ και ολοκληρώσαμε το θέμα του Θιβέτ. Ακολουθεί τώρα το θέμα του μέλλοντος της πράξης για την ενιαία αγορά. Ξεκινά ο συνάδελφος Στάντλερ. Ευχαριστώ. Ήδη έχω πει ότι θα ψηφίσω κατά αυτού του ψηφίσματος ε, που είναι σαν εικονικό φάρμακο. Βλέποντας ε, ε, τον κατάλογο του, που έπαιξε ο Άλεν Γκρίνσπαν και τα όσα είπε η κυρία Λαγκάρντ, είπε ο Γκρίνσπαν ότι έχει αποτύχει το, το ευρώ και τώρα απειλεί να καταστρέψει και την εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ε, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα ε, είναι ένα ψήφισμα που είναι σαν εικονικό φάρμακο, ψευδοφάρμακο για την ε, ενιαία αγορά και θα δυσκολέψουμε ακόμη περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να, να επιζήσουν και να μπουν στο σωστό δρόμο. Επικροτούμε τη γραφειοκρατία, θα έπρεπε να την διαλύσουμε γιατί πνίγει τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει. Δεν δημιουργούμε θέσει απασχόληση κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε με πολιτικέ αποφάσει, αλλά θα πρέπει με συγκεκριμένα μέτρα να προωθήσουμε τι ε, θέσει απασχόληση. Γι' αυτό σα λέω ότι αυτό το ψήφισμα είναι εικονικό φάρμακο, ψευδοφάρμακο και το καταψήφισα. Ευχαριστώ κύριε Στάντλερ. Κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν συμμερίζομαι την τοποθέτηση του προηγούμενου συναδέλφου. Θεωρώ ότι το κοινοβούλιο αυτό πολύ καλά άσκησε τα δικαιώματά του και τις αρμοδότητές του εγκρίνοντας το ψήφισμα αυτό που ψηφίσαμε. Είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να συμπληρωθεί η οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς χωρίς να προσθέθούν νέοι νόμοι, αλλά υλοποιώντα τη δέσμη μέτρων, νομοθετικών μέτρων που έχουμε στα χέρια μας. Ε, ανάπτυξη τη ενία αγορά θα πρέπει να λάβει υπόψη τέσσερι βασικέ συνιστώσει που περιέχει το ψήφισμα αυτό. Τη διάσταση των εργαζομένων, διότι πάνω από το 90% τη αγορά μα ανήκει στην δράση και οφείλεται στη δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίση, στην κοινωνική αξία των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να ε, ε, σταθμίσουμε και πάλι του κανόνε μα ε, προ όφελο των πολιτών. Την ε, διατομιακότητα τη αγορά, τον οριζόντιο χαρακτήρα τη και τέλο τον την ε, τάση να πολλαπλασιάζονται οι συνέπειες από την αγορά σε εθνικό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να κάνω και την εξή παρατήρηση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που εγκρίθηκε η τροπολογία εκτός μικροφωνών μιλητρία. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Ματσόνη. Συνάδελφος Νικολάη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της εκθέσεως αυτής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Έτσι αποκτούμε όραμα και έχουμε και λύσεις γιατί πρόκειται για πυλώνα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Πρόκειται λύσεις και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας την οποία εάν μειώσουμε κατά 25% μέχρι το 2015 θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό στόχο. Θα πρέπει να και τα κρατη Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν ό,τι μπορούν. Και τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι εταιρείε έτσι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα. Θα πρέπει να έχουμε επίση για να αμοιβή αναγνώριση ε, των επαγγελματικών προσόντων όπως προβλέπει το άρθρο 59 της οδηγίας. Και έτσι θα ε, βελτιωθεί και παραργασία. Ευχαριστούμε την κυρία Νικολάη. Η κυρία Ρόιτοβα δεν είναι παρόν, ε, παρούσα. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά ψήφισα υπέρ αυτό του σημαντικότατου, αυτή τη σημαντικότατη έκθεση. Εκτός από το άρθρο 22, όπου γίνεται λόγος για το συντονισμό των φορολογικών πολιτικών. Δεν συμφωνούμε, ή μάλλον έχουμε ενδιασμούς ω προ το σημείο αυτό. Αυτό δεν μας επέτρεψε να υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο εντάφιο. γι' αυτό και απήχαμε. Πέραν αυτού, είναι πολύ καλές παρατηρήσεις που γίνονται σε αυτή την έκθεση. Και αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την ενιαία αγορά, τουλάχιστον θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από την οικονομική κρίση. Δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέλλη. Κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, υπερψήφισα το, το, έκδοση ναι, αυτή, διότι η νέα αγορά είναι ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είναι σημαντικό για την πορεία τη ενοποίησης. Υπάρχουν πολλέ προκλήσει που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τόσα πολλά που ακόμη απομένει να επιτευχθούν από την ενιαία αγορά. Είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να στηρίξει την οικονομία και να δημιουργήσει νέε θέσει εργασία. Από αυτή την άποψη, νομίζω η νέα αγορά θα πρέπει να είναι κάτι που θα απασχολήσει περισσότερο τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε ευφυή βιώσιμη ανάπτυξη που να προωθεί την ε, συμμετοχή και εδώ θα πρέπει να λεφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Χρειαζόμαστε περισσότερη κινητικότητα των ε, επαγγελματιών με προσόντα, των εργαζομένων με προσόντα, ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι πιο ανταγωνιστική. Νομίζω ότι η εξακολούθηση των ε, περιορισμών που έχουν επιβληθεί στους Ρωμανούς εργαζομένους πρέπει να έρθουν. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Καμάλ έχει το λόγο. Ένα από τα λυπηρά θέματα από την αντίθεση δράση πολλών ε, μελών εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι παρότι και πολλών πολιτικών παρότι διαμαρτύρονται για τη λιτότητα δεν έχουν ε, κάποιο πρόγραμμα για να την ε, αναστείλουν. Η λιτότητα σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία διαθέτουμε και παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνουμε αναπτυξιακά μέτρα για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε πιστεύει κανείς είτε όχι στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ενιαία αγορά και καλωσορίζω τις προτάσεις για το μέλλον της ενιαίας αγοράς που θα μειώσουν τα σύνορα μεταξύ κρατών μελών ε, και θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του προστατευτισμού. Ας δώσουμε μεγαλύτερη αγορά και μεγαλύτερο περιθώριο στις εταιρείε να έχουν μια μεγαλύτερη πλατφόρμα για να μπορέσουν ε, να κάνουν εμπόριο με την Ευρώπη και όχι με άλλες χώρες στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμάλ, ο συνάδελφος Τάνοκ. Ψήφισα υπέρ, Πρόεδρε, όσον αφορά αυτό το ψήφισμα για την ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα λίγα καλά που έχουμε εδώ πέρα στην αγορά έχουν ωφελθεί πάρα πολύ, ευκαιρίε για τι επιχειρήσει, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Στη σημερινή συγκυρία τη κρίση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ό,τι μέτρα παίρνει η Ευρωζώνη για μια ένωση τραπεζική δεν θα πρέπει να παγώσει τον τομέα ε, αυτών ε, της, της γιατί το, το, το του Λονδίνου είναι η εκλογική περιφέρεια και περήφανος γι' αυτό και τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε σημαντική νομοθεσία και γρήγορα και έτσι να είμαστε πιο ε, αποτελεσματικοί όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, να μην έχουμε άλλη γραφειοκρατία και οι θεμελιώδεις ελευθερίες διακίνησης να αναβαθμιστούν. Ευχαριστούμε κύριε Ντάνοκ. Ολοκληρώσαμε τις επεξηγήσεις ψήφου για το μέλλον της πράξης για την αγορά. Ακολουθούν οι επεξηγήσεις για την πρώτη ψηφίσματος μέλλον του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου. Η συνάδελφος Ματσόνη. Και πάλι ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δοθεί μια κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ακριβώ για να δοθεί και μια σωστή κατεύθυνση στι δημόσιε διαβουλεύσει για το μέλλον του εταιρικού δικαίου στην Ευρώπη. Όπω προκύπτουν τα δεδομένα που έχουμε από μελέτε, που περιλαμβάνει και η έκθεση αυτή, περισσότερε εταιρείε και επιχειρήσει λειτουργούν εντό ε, νέα αγορά, αλλά με διασυνοριακά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ενοποιηθούν τα εταιρικά πρότυπα και τα μοντέλα των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει τις κατάλληλες ε, τα κατάλληλα συνθήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει, δηλαδή την εναρμόνιση, την ομογενοποίηση, την πρόθεση της κινητικότητας, τη διαφάνεια. Ελπίζω η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει εν το χρόνο, ιδίως μετά την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε την κυρία Ματσόνη. Η κυρία Ρόιτοβα πάλι δεν είναι εδώ. Συνάδελφος Μπίλαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολλά τα μέτρα που σκοπό έχουν να προωθήσουν τη διαφάνεια και να πλουστεύσουν τους ε, κανόνες στις επιχειρήσεις και τις εμπορικές τους σχέσεις. Είναι καλά τα νέα για τις επιχειρήσεις και θα επιτρέψει να αναθερμανθεί ο ανταγωνισμό στην αγορά, το εταιρικό δίκαιο και η πλουστεύση του. Επίσης, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα που ακριβώς προκύπτουν λόγω της διαφορετικής ερμηνεία του δικαίου. Είμαι υπέρ λοιπόν και ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος της έκθεσης ακριβώς γιατί είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες απλούστευσης για το επιχειρησιακό περιβάλλον και για τον περιορισμό του γραφειοκρατικού άχθους. Επίσης, εδώ έχουμε να κάνουμε και με κοινού κανόνες και να διαφανέστερο σύστημα οικοδόμησης των σχέσεων ιδιοκτησίας. Η Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία επίση είναι κάτι που και πάλι θα ωφελήσει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ τη έκθεση αυτή του ψηφίσματος, δηλαδή της πρότασης ψηφίσματος, διότι το εταιρικό δίκαιο είναι καθοριστικής σημασίας από την πλευρά της ε, λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Είναι απαραίτητο ε, για την προάσπιση των ε, εταιριών και των δικαιωμάτων τους και για λόγους νομικής βεβαιότητας. Χρειάζεται λοιπόν ένα επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να ακολουθεί τους ρυθμούς των εξελίξεων γύρω μας. Μεταξύ άλλων λοιπόν, επικαιροποίηση του εταιρικού δικαίου, ναι, είναι ανάγκη αυτό προς όφελος των μετόχων και των ε, πελατών των εταιριών. Θα ήθελα εδώ να τονίσω το ρόλο των ε, διαφόρων εταιριών στην προσφορά τους, συμβολή τους, στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Περισσότερα θα πρέπει να γίνουν στον ε, τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επίσης. Το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν απλούστερη πρόσβαση στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσαν οι επεξηγήσει ψήφου για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου και ακολουθούν οι επεξηγήσει ψήφου για την πρόταση ψηφίσματο στοχεύοντα σε μια ανάκαμψη με άφθονε θέσει απασχόληση. Η κυρία Ματσόνη έφυγε. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σήμερα ημέρα τέτοιες ε, αναλύσεις, τέτοιες εκθέσεις θεωρούμε ότι αποτελούν πάρα πολύ σημαντική συμβολή στην πολιτική μας ε, διότι εδώ έχουμε πάρα πολύ σωστή προσέγγιση όσον αφορά την αγορά εργασίας στην Ευρώπη διότι να θέλω να σας αναφέρω αυτά που αναφέρω εδώ η έκθεση για το ότι δεν έχουμε συνδυάσει ε, το πανεπιστήμιο με την ε, με την πραγματικότητα στην αγορά γιατί δεν έχουμε αρκετούς μηχανικούς, δεν έχουμε αρκετούς τεχνικούς. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση που πρέπει να είναι διαρκής. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουμε την φορολόγηση της εργασίας τόσο όσο το κάνουμε σήμερα σε τόσα Επίσης θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντικό βήμα. Είναι μια έκθεση πάρα πολύ ενεργητική που θα πρέπει να τη λάβουμε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Κύριος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης. Από το Υπουργείο Αλήθειας του Όρουελ προέρχεται αυτή η φράση και δεν θα σας κουράσω άλλο με τον Όρουελ σήμερα. Θυμάμαι την ατζέντα της Λισαβόνα όταν πρώτο ήρθα στο Κοινοβούλιο. Το θυμάστε, θα έδινε στην Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο μέχρι το 2010. Πάει το 2010, ήρθε και έφυγε. Και θα μας έλεγε κανείς, ε, μα τι κάνατε. Μετά άρχισαμε να λέμε για το ευρώ και λέγαμε διάφορα επιχειρήματα για την ε, Οικονομική Νομισματική Ένωση. Πώς θα πάμε όλα αυτά. Και τώρα για το τελευταίο δείγμα ύβρεο, ε, οι πολιτικοί. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση, ακόμη και αν απασχολώ κάποιον ε, στο γραφείο μου. Το κάνω με χρήματα των φορολογουμένων που τα παίρνουν από τον ιδιωτικό τομέα που θα τα χρησιμοποιούσαν ε, με μεγαλύτερη επιτυχία. Καταστρέφουμε θέσει απασχόληση. Θα πρέπει να δώσουμε στου επιχειρηματίε που είναι πραγματικά η ατμομηχανή τη οικονομία, να δημιουργήσουν πραγματικέ θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χάναν. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Χάναν ότι είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένο ο τίτλος και όταν χρησιμοποιούμε ένα τόσο εμπνευσμένο τίτλο θα πρέπει να ανταποκρίνεται και το περιεχόμενο και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν σημαντικό το ότι σήμερα το πρωί ψηφίσαμε υπέρ ενός πακέτου επενδύσεων για να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Αυτό δίνει ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ότι πραγματικά προσπαθούμε να επανισορροπήσουμε τη λιτότητα με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης και ελπίζω να τα ακούει το Συμβούλιο και να τα σημειώνει και να λαμβάνει δράση. Και όταν οι Ιρλανδοί πολίτες ψήφισαν υπέρ του Δημοσιονομικού Συμφώνου, περίμεναν τέτοιε επενδύσεις σαν κομμάτι του πακέτου. Είναι δύσκολε. είναι ε, περιορισμένε οι δυνατότητε που έχουμε για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόληση. και ένα τομέα είναι η κατάρτιση των εργαζομένων, γιατί εκεί υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο να αποσύρει ε, την δεσμευτική μειοψηφία για το Ταμείο παγκοσμιοποίηση και να μα αφήσει τη δυνατότητα του Ταμείου παγκοσμιοποίηση για την κατάρτιση των ε, απολυθέντων. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Συνάδελφος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, δεν ναι, έκανα μικρό λάθος ότι είναι ψηφοφορίες. Γιατί? Γιατί στην πρώτη ψηφοφορία πάτησα το λάθος κουμπί. Θα ε, μιλήσω με τους ε, αρμοδίους γι' αυτό. Και έχουμε πει ότι είπαμε 80-85% τωρα ε, Τώρα έχουμε 68-69%. Και αυτό σημαίνει 17 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πρέπει να ανακτήσουμε. Καλά έλεγες ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε θέσεις εργασίας εμείς οι ίδιοι, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις, τις, ε, πιο κατάλληλες συνθήκες προς τούτο. Και σας παραπέμπω σε αυτό που είπε ο Επίτροπος Μπάρνιε ηλεκτρονικό εμπόριο, ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία, όλα αυτά μαζί, εάν τα προωθήσουμε, μπορούν να βοηθήσουν. Και έτσι το 2020 έχουμε φτάσει στο 75% απάσχολη στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Κυρία Μπαθέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι συμφωνώ η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα δημιουργηθούν και θέσει απασχόληση. Πολλοί άριθμε συζητήσει έχουν γίνει για το ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προτάσει, το Συμβούλιο έχει λάβει αποφάσει. Τώρα πρέπει να υλοποιηθούν με συγκεκριμένε χειροπιαστέ ενέργειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι σαφή και ανένδοτη για τα 82 εκατομμύρια ευρώ, δις ευρώ μάλλον, για το πώ θα δαπανηθούν για θέσει εργασία για του νέου προκειμένου να προωθηθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για τους νέους επιχειρηματίες. Έχω θέσει και ερώτηση, απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Και εκφράζω την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει και για τους νεαρούς επιχειρηματίες ως το τέλος της φετινής χρονιάς. Πρέπει κάτι να γίνει ώστε να ε, προλύνεται το έδαφος για να μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν στην ε, ενιαία αγορά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό και φάνηκαν οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των αριστερών που πιστεύουν στην παρέμβαση του κράτους και των δεξιών που πιστεύουν στην, ε, στον φιλελευθερισμό και της αριστεράς πιστεύουν ότι με τη χρήση των ε, εισοδημάτων των φορολογουμένων θα δημιουργήσουν τεχνητέ θέσει εργασία. Όμω θα φορτώσουν και άλλο στην κοινωνική πρόνοια. Και όταν φτάνουν στι εκλογέ, του λένε αν ψηφίσετε τα κόμματα τη δεξιά, όχι μόνο θα χάσετε τη θέση εργασία σα, αλλά και τα επιδόματά σα. Ενώ όσοι είναι στη δεξιά πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να γίνει να δημιουργηθούν οι κατάλληλε προποθέσει για ανάπτυξη. Να φεύγει η κυβέρνηση ε, ε, από το δρόμο της αγοράς των επιχειρηματιών, να τους επιτρέπουν να δημιουργούν νέες θέσει και μάλιστα βιώσιμες, όχι που να εξαρτώνται από τις δαπάνες ε, του κράτους, να είναι βιώσιμες στον ιδιωτικό τομέα και όλοι να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καμάλ. Ολοκληρώσαμε τις επεξήγησεις ψήφου για το, την πρόταση ψηφίσματος για την ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης και ακολουθούν οι επεξήγησεις ψήφου για, τις για την πρώτη ψηφίσματος για του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων γυναικών. Η κυρία Ματσόνη δυστυχώ χρειάστηκε να φύγει και θα αρχίσει η κυρία Νικολάη. Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματο για δύο λόγου. Δυστυχώ, μέσα στον 21ο αιώνα ακόμη έχουμε τέτοιου είδου βάρβαρες πρακτικές, αυτές τις βίες πρακτικές κατά των γυναικών. Ακόμα συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πολλές φορές για θρησκευτικού λόγους, 500.000 γυναίκες στην Ευρώπη μόνο υφίστανται τους αγροτηριασμούς. Θα πρέπει επομένω τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν δράση και αυτό το φαινόμενο δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί, να εξαπλωθεί στην Ευρώπη είναι άσχετο παντελώ με ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτισμένη συμπεριφορά. Πάρα πολύ ε, πρέπει να προστίξουμε αυτή την έκθεση. Είναι ένα καμπανάκι. Κυρία Ζαμπόσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο Οργανό Υγεία λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 500.000 γυναίκε ανήλικες και ανήλικε που έχουν υποστεί εκδοτηρισμό γενετικών οργάνων. Και άλλε 180.000 απειλούνται να υποστούν τον εκδοτηρισμό. Πρόκειται για αποτρόπια πρακτική. Δεν έχει σχέση με καμία θρησκεία. Είναι μια παράδοση που όμως έχει ισοπεδωτικό αποτέλεσμα για τις ζωές των γυναικών. Είναι το δεύτερο ψήφισμα που έχουμε για αυτό το θέμα που καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη κάτι να κάνουν για να σταματήσει κάτι τέτοιο και ποτέ νομίζω ότι πολλά μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτό το βίο φαινόμενο γιατί έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τις οργανώσει εκείνε, ε, οι οποίε βοηθούν τα θύματα και επίση στο πλαίσιο μια τέτοια προσπάθεια αλλαγή μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ε, αποφασιστικά ούτω ώστε να σταματήσει μια τέτοια αποτρόπια πρακτική. Ζάβε, ευχαριστώ. Μπασέσκου. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, διότι ο κριτηριασμός γενετικών οργάνων είναι απαράδεκτος, είναι βαρβαρότητα. Είναι μια σωματική και ψυχολογική βία που ασκείται στις γυναίκες με τεράστιες συνέπειες θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρότατες επιπλοκές στην υγεία ή και στο θάνατο. Είναι μάλιστα παράνομη πρακτική αυτή, αλλά ακόμη μπορεί να ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τουλάχιστον 3 εκατομμύρια γυναίκες να υποφέρουν στην Ευρώπη, ακόμη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω υπόψη μια συγκεκριμένη περίπτωση σε μια γνωστή οικογένεια όπου τέσσερα κορίτσια υποβλήθηκαν σε ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων. Ελπίζω ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα εγκρίνει το σχετικό ψήφισμα για το θέμα αυτό. Η ενημέρωση για τους κινδύνους και τις επιπλοκές είναι τεράστια σημασία. Ευχαριστούμε κύριε Μπασέσκου. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματο ε, για τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων γυναικών. Ε, εκτιμάται ότι 100 ε, εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών ζουν κάτω από τον κίνδυνο τέτοιων ακροτηριασμών. Στο κέρας της Αφρικής είναι παραδοσιακή πρακτική, αλλά δεν είναι απέτηση καμιάς θρησκείας. Είναι μια βάρβαρη πρακτική κορίτσια κάτω των 15 ετών ε, ζουν ε, με μακροπρόθεσμες ε, δυσμενείς συνθήκες με πάρα πολλές συνέπειες όπως αιμορραγίες, μολύνσεις, ακόμη και από τον ιό του AIDS. Και μπορεί να είναι και μοιραίες αυτές οι πρακτικές. Ευχαριστούμε και από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να απαγορευτεί σε όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών και να ποινικοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται δίωξη και των γιατρών και των ε, γονέων που καταφεύγουν σε αυτήν την πρακτική. Για λόγους πολιτισμικής ε, ε, Ιδιαίτεροτητα η αστυνομία πολύ συχνά δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε και Ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσει ψήφου για το θέμα αυτό και περνάμε στι επεξηγήσει για, το για την τελευταία πρόταση ψηφίσματο. Οι συνάδελφοι Ζουιβάν, Χάρκιν δεν ήταν και Ματσόνη δεν είναι παρόντε. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το σκάνδαλο των εμφυτευμάτων στήθους είναι ένα παράδειγμα ε, ανικανότητας και νομοθετικών ε, κενών. Ελπίζω ότι ε, η Επιτροπή τώρα θα προσπαθήσει να θεσπίσει το κατάλληλο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα εμφυτεύματα στήθους και για τα ιατρικά προϊόντα ώστε να καλύπτεται όλη η αλυσίδα της παραγωγής και της εμπορίας και να ενδυναμώσει την παρακολούθηση της αγοράς από τα κράτη-μέλη. Ως γιατρός χαιρετίζω το ψήφισμα αυτό. Χρειάζεται ένα σύστημα ταυτοποίησης, ούτως ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα των εμφυτευμάτων στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζαμπόσκα. Τελειώσαμε λοιπόν με τις επεξηγήσεις ψήφου και για τα ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους. Τελειώσαμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ζαμπόσκα, τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του Διερμήνης και διακόπτη τη συνεδρίαση.